Ε, να εγκρίνουμε την μέσα διάταξη αν δεν έχετε αντίρρηση και για την διερμηνία να σας ενημερώσω ότι ακολουθούμε την πλατφόρμα ε, Interaction 2 και οι γλώσσες που μπορείτε να μιλήσετε είναι η συνήθιση μαζί με τσεχικά και σλοβενικά και το απόγευμα δεν θα έχουμε σλοβενικά και ε, λιθουανικά καθώς και σλοβενικά και τσεχικά. Παρακαλώ όταν ε, μιλάτε, όταν δεν μιλάτε, να κλείνετε το speak ε, και όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση μπορείτε μέσω διαδικτύου. Για τους εξαποστάσεως συμμετέχοντες μπορείτε να ε, κλείνετε τη σύνδεσή σας όταν δεν θέλετε να συμμετάσχετε από τις 2 παρατέταρτο έως τις ε, Τρει παρατέταρτο θα έχουμε την πρώτη σύνοδο ψηφοφοριών, ο πρώτος γύρος και τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν μέσω email. Ο δεύτερος γύρος, τελική ψηφοφορία, θα λάβει χώρα μετά τις ανακοινώσει των αποτελεσμάτων μέσω email. Είναι σημαντικό να είστε εδώ ε, προσωπικώ ή να συνδεθείτε στη συνεδρίαση Apple πριν τον πρώτο γύρο των ψηφοφοριών. Δύο παρατέταρτο διότι θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει απαρτία, δηλαδή 40 μέλη. Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 3 και 4 της σας διάταξης που θα συζητήσουμε. Πρέπει να πω ότι καλωσορίζω την συζήτηση που θα κάνουμε και χαίρομαι για αυτή, διότι θεωρώ ότι το να έχουμε επίκαιρα και εύστοχα στατιστικά δεδομένα και δείκτες είναι πολύ σημαντικό για να καταπολεμήσουμε την ένδια και τι ανισότητε, για να βελτιώσουμε την ένταξη των πολιτών και την καλύτερη στόχευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, να εντοπίσουμε τα ε, ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες των πολιτικών μα και να τι βελτιώσουμε. Για όλου αυτού του λόγου. χρειαζόμαστε δεδομένα. Ε, γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που εγκρίνονται το πλαίσιο των κοινωνικών στατιστικών στοιχείων, όπως σχεδιάστηκε πέρσι, μετά από τις επικοδομητικές μας διαπραγματεύσεις. Και ολοκληρωμένο, το ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικών στατιστικών, όπου το Κοινοβούλιο έχει ε, σημαντικό λόγο για τον καθορισμό των μεταβλητών. Τα σχετικά δεδομένα θα συλλέγονται στα κράτη-μέλη, ανάλογα με τις πολιτικές ανάγκες, και θα εξυπηρετήσουν πάρα πολύ τη δουλειά μας για την ε, ε, υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα, του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Σήμερα θα συζητήσουμε τις καταξιοσοδότηση πράξεις για σημαντικά δεδομένα, για το ICT, για τις εργασιακές δεξιότητες και τα σχετικά δεδομένα για τους συνταξιούχους. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα όλα. Θα δώσω τώρα το λόγο τον ε, κύριο Μεσιντιακλίν ε, της Eurostat, διευθυντή της Eurostat, για μια σημαντική παρουσίαση. Και μετά στους συναδέλφους του για να συμπληρώσουν. Κύριε Μερσή, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σε αυτή την ε, εξαποστάσεως συνεδρίαση για να μιλήσω για αυτή τη σημαντική κατεξοδότηση πράξη. Μ' ακούτε σωστά. Ναι, σας ακούμε και σας βλέπουμε. Όλα είναι εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ. Τα πράγματα έχουν ως εξή. Στρεφόμαστε ξανά προς εσάς για μια επιπλέον κατεξοδότηση πράξη, διότι όπως είπατε πολύ σωστά, απαιτούνται περί σώτερα δεδομένα για τα κοινωνικά θέματα. Στην ε, προκειμένη περίπτωση για την απασχόληση, της συνθήκες διαβίωσης, αλλά και για την υγεία, την παιδεία και άλλους ε, τομείς της ζωής των πολιτών. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται σε διάφορες ε, περιπτώσεις. Η σημαντικότερη είναι το πίνακας αποτελεσμάτων των δικτών που άπτεται του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Το εξάμεινο στο οποίο χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο δεδομένα για κοινωνικά θέματα. Φυσικά σε τέτοιες εποχές κρίσης κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο ώστε να προσπαθήσουμε να παρακολουθούμε και να βοηθάμε την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής και έτσι τα δεδομένα αυτά που ζητάμε χρειάζονται για να αξιολογούμε, να διατυπώνουμε, να παρακολουθούμε και να εξετάζουμε τις επιπτώσεις των πολιτικών που χαράσσονται. Έχει διαπιστωθεί η ανάγκη ανανέωσης της υποδομής ε, της στατιστικής, διότι την τελευταία 20 αιτία οικοδομήθηκε βήμα προς βήμα αλλά σιγά σιγά φτάνουμε στα όρια του τι είναι δυνατόν με, τα με το σημερινό πλαίσιο για τον λόγο αυτό. Ε, γι' αυτό προτείνουμε ανανέωση αυτού του κανονισμού 19700 ΓΕΣ που περιλαμβάνει τα ολοκληρωμένα στατιστικά ε, στοιχεία και γι' αυτό τον κανονισμό είχαμε ε, σοβαρή υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον 219.700 και εκφράστηκε και η επιθυμία να συμμετέχει το Κοινοβούλιο σε βάθος και ένεργα σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας. Αυτός ο κανονισμός πλαίσιο περιλαμβάνει 7 ε, δράσεις συγκέντρωσης δεδομένων αφορούν την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης, τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, ε, την υγεία, την παιδεία, την κατανάλωση και την έρευνα. Τι θέλουμε να κάνουμε με αυτό το νέο κανονισμό, να υποστηρίξουμε καλύτερα την ε, δημιουργία πολιτικών, περιλαμβάνοντας περισσότερα θέματα, τα οποία θα βοηθούν περισσότερο στη χαράξη πολιτικής. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε την ποιότητα των δεδομένων που παρέχουμε, ειδικότερα θέλουμε να παρέχουμε αυτά τα δεδομένα πιο έγκαιρα και πιο επίκαιρα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα το τομέα των συνθήκων διαβίωσης. Από πιο τεχνική άποψη τώρα υπάρχουν διάφορες βελτιώσεις. Έχουμε απλουστεύσει την συγκέντρωση δεδομένων, την έχουμε χωρίσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες ώστε να ε, συγκεντρώνονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο και κάνουμε καλύτερη ανάλυση σε σχέση με το παρελθόν λόγω της ομοδοποίησης που έχουμε εφαρμόσει. Έτσι λοιπόν ε, Γι' αυτό το λόγο θέλαμε σήμερα να έχουμε έναν κανονισμό πιο ευέλικτο. Ένα από τα προβλήματα από τον προηγούμενο κανονισμό ήταν η δυσκολία προσαρμογής σε νέε συνθήκε. Σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θέλαμε λοιπόν ο κανονισμός αυτός ε, να γίνει πιο ευέλικτος. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω κατεξουδότηση πράξεων. Η καταξιοδότηση πράξης ε, που προβλέπονται αφορούν ε, τρεις ε, τομείς. Πρώτον το σχεδιασμό, που βασίζεται στην πρόβλεψη του τι μπορεί ή θα συγκεντρωθεί ως στοιχείο μέσα στα επόμενα χρόνια με κάποια δυνατότητα φυσικά ευελιξίας και προσαρμογής, τα θέματα τα οποία ενδεχομένως θα καλύπτονται, τα οποία ορίζονται στη νομική βάση, αλλά μπορούν να διευρυνθούν και να προσαρμοστούν σε κατεξούδαση πρέπει και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ο αριθμός και ο τίτλος των μεταβλητών που θα συμπεριληφθούν σε κάθε συγκέντρωση δεδομένων που δίνει στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να εξετάζει και να σχολιάζει και να εκφέρει άποψη ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο για το εκάστοτε ζήτημα. Σήμερα λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά που ζητάμε μια κατεξουδότηση πράξη. Κάποιες βασικές ε, κατεξουδότηση πράξεις ε, εγκρίθηκαν ήδη πέρυσι, αυτές που ήταν ε, πιο επίγουσες. και που αντιστοιχούσαν ε, στο επίκεντρο του τομέα των συνθήκων διαβίωσης και του επίκεντρο του τομέα ε, του εργατικού δυναμικού. Εδώ λοιπόν σας παρουσιάζουμε το πυρήνα των ICT, των τεχνολογιών ε, πληροφορίας και επικοινωνιών. Είναι ένας ιδιαίτερος τομέας απαιτεί ταχεία εξέλιξη. Εξελίσσεται πολύ γρήγορα από μόνος του. Και το χρονικό πλαίσιο για την υιοθέτηση αυτού του συγκεκριμένου θέματος που αλλάζει, μεταβάλλεται κάθε χρόνο, έχει κάπως προσαρμοστεί στον κανονισμό. Σήμερα επίσης έχουμε και κάποια τμήματα. Δεν είναι το κεντρικό κομμάτι της έρευνας ε, για το εργατικό δυναμικό, αλλά κάποια επιπλέον ε, τμήματα τα οποία θα αφορούν το μέλλον. Αποτελούν κομμάτι του μηχανισμού που έχει ενσωματωθεί θεσπιστεί από τον κανονισμό ώστε να βελτιωθεί η ευελιξία. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτή ήταν η γενική μου εισαγωγή. Θα μπορούσαμε να περάσουμε σε ένα από τα δύο θέματα ενδεχομένω. Ναι, ευχαριστώ. Thank you. Thank you. Ναι, ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κράλ η οποία θα παρέμβει για το σημείο 3 αν δεν κάνω λάθος. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους θα παρουσιάσω τον κανονισμό για τη συλλογή των τίτλων και των αριθμών διαφόρων ε, ε, προϊόντων νέων τεχνολογιών ε, για το 2021. Ο κανονισμός θα μας επιτρέψει να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία για πολιτικές που έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση, παραδείγματος χάρη θα χρησιμοποιηθεί στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, θα υπάρξουν δείκτες για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, τα, ψηφια, τα ψηφιακές δεξιότητες, μεταξύ άλλων. Και αυτό θα γίνει σαν οικοκυριά, αλλά και σε άτομα, για άτομα 16 74 ετών, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, θα πρέπει να έχουμε μία μελέτη κάθε χρόνο και να την προσαρμόζουμε και εδώ για το 2021 έχει γίνει μια προπαρασκευή από κοινού με τους ειδικούς στατιστικολόγους των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών. Ε, υπάρχουν task force, ομάδες εργασίας και ταυτόχρονα ε, λαμβάνουμε υπόψη τις ε, ανάγκες του χρήστη αλλά και τις πολιτικές ανάγκες για το 2021 εξετάζουμε και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ψηφιακές δεξιότητες... αλλά και την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες καθώς και η συχνότητα της χρήσης τους, οι δραστηριότητε στο ίντερνετ, αλλά και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα προβλήματα, ε, τα όρια της, ε, των νέων τεχνολογιών και τα θέματα ιδιωτικής ζωής και προστασίας της. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύντομη εισαγωγή και τώρα τον λόγο έχει η κυρία Αν Φερμάνς. Όχι, η Αν Κλεμονσόν παρακαλώ, η οποία θα μας μιλήσει για το σημείο 4 που ασχολείται με τα ζητήματα ψηφιακής αγοράς και ε, διαβίου μάθησης. Παρακαλώ. Δεν είναι συνδεμένη. Μάλιστα, ο κύριος Μέρση έχει το λόγο, παρακαλώ. Ναι, φαίνεται να υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Η κυρία Κλεμονσό ε, τη ζητούν ε, ε, κάποιο password για να μπορέσει να συνδεθεί. Δεν ξέρω αν μπορείτε αυτό να το ε, λύσετε το ζήτημα. Έχουμε χάσει την επαφή με την κυρία Κλεμόνσο. Σας βλέπουμε τώρα κυρία Κλεμονσό. So Anne Clemenceau has a Δυσκολεύεται να συνδεθεί η κυρία Κλεμόνσο. Οπότε αν δεν έχετε αντίρρηση κυρία Πρόεδρε, θα αυτοσχεδιάσω κάπως και θα κάνω εγώ την παρουσίαση αν δεν έχετε αντίρρηση. Ναι βεβαίως κύριε Μέρση. Ναι, συγγνώμη γι' αυτό. Όπως είπα, σε ό,τι αφορά το LFS, την ε, έρευνα δηλαδή για την αγορά, για την για το εργατικό δυναμικό υπάρχει μια ευελιξία στον κανονισμό. Έχουμε τον πυρήνα του ελεφές της μελέτης αυτής, οι ερωτήσεις και μεταβλητές που συλλέγουμε κάθε χρόνο και που έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό με τα πιο βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με, το, με την απασχόληση και που συμπληρώνονται κάθε χρόνο με επιπλέον μεταβλητές ε, οι οποίες συναλλάσσονται. Γιατί συμβαίνει αυτό. Θέλουμε να επιτρέψουμε να βρεθεί χώρος μια και έχουν περιορισμούς σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να συλλέξουμε όλες τις μεταβλητές κάθε χρόνο. Πρέπει να βρούμε λοιπόν λύσεις έτσι ώστε να έχουμε ε, έναν λογικό, ένα λογικό χρονικό διάστημα για αυτήν την συνέντευξη, να μην ξεπερνάει κάποια όρια χρονικά δηλαδή. Και κάποιες ερωτήσεις λοιπόν ε, τις θέτουμε κάθε 8 χρόνια ας πούμε κάθε 2 χρόνια που δεν είναι οι πιο σημαντικές. Έχουμε την τακτική ε, συλλογή δεδομένων που συλλέγουμε κάθε χρόνο και κάποια ζητήματα ad hoc τα οποία, για τα οποία συλλέγουμε στοιχεία κάθε τέσσερα χρόνια ας πούμε. Ad hoc ζητήματα που αποφασίζονται με βάση την ε, τρέχουσα κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα την πράξη κατεξιοδότηση που περιλαμβάνεται εδώ στο πακέτο Μιλάμε για το 2022-2023 και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, συμμετοχή στην αγορά εργασίας και τα job skills. Ε, πρόκειται για ένα διαφορετικό ζήτημα τα job skills και από εκεί πέρα, δηλαδή είναι ad hoc ζήτημα και από εκεί πέρα έχουμε ε, το ε, πιο τακτικό ζήτημα των ε, συντάξεων και της αγοράς εργασίας. Το θέμα των job skills το συντονίζουμε με άλλες διεθνείς οργανώσεις, το θέμα των δεξιοτήτων εργασίας. Είναι ένα σημαντικό θέμα, το συντονίζουμε με τον ΩΣΑ, στα πλαίσια πιο συγκεκριμένα του ΠΙΑΚ και με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα, το Eurofund, που ασχολείται με τις μελέτες για τις ευρωπαϊκές συνθήκες εργασίας. Το νόημα αυτού του τμήματος, αυτού του module, είναι να εντοπίσουμε στοιχεία για την απασχόληση που αλλάζουν με βάση την τεχνολογική πρόοδο και να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση με βάση τα προφίλ των διαφόρων δεξιοτήτων, των διαφόρων καθηκόντων και να εξετάσουμε διάφορα, τα διάφορα καθήκοντα που συνδέονται με τις διάφορες θέσεις απασχόλησης. Εδώ ο, ο στόχος είναι τα άτομα 15-74 που εργάζονται αυτή τη στιγμή ή που εργάστηκαν στους τελευταίους 24 μήνες και το module αυτό, το τμήμα αυτό βασίζεται στην κατηγοριοποίηση των καθηκόντων με βάση δύο διαστάσεις. Το περιεχόμενο των καθηκόντων αυτών καθ' αυτών, δηλαδή τι κάνουν τα άτομα αυτά στο χώρο εργασία τους και τα, οι μέθοδοι και, εργαλεία, και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να υλοποιηθούν αυτά τα καθήκοντα. Το πώς δηλαδή δουλεύουν, τι κάνουν και πώς εργάζονται. Το Module 2023, το επόμενο δηλαδή για την ε, για τη συντάξη και τη συμμετοχή στην αγορά εργασία έχει ω πληθυσμό στόχο τα άτομα από 50 έω 74 και βασιζόμαστε στα πρώτα στοιχεία ε, τα συνταξιδοτικά. Δεν βασιζόμαστε στους ανθρώπους δηλαδή που ε, εργάζονται, που είναι στην αγορά εργασίας, Μιλάμε για τη μετάβαση από την αγορά εργασίας προς την συνταξιοδότηση. Επικεντρωνόμαστε δηλαδή ε, σε αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Μερσή να ακούσουμε τους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο για τα θέματα αυτά. Πρώτος ο κύριος Κώσα από το ΕΛΚ. Δύο λεπτά για το κάθε μέλος. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον διευθυντή που είναι εδώ. Είναι παλιός ε, γνωστός, παλιός φίλος. Γιατί μου σκιώδησε συγκεκριτής εκ μέρους του ΕΛΚ όταν, συζητούσαν τον, συζητούσαμε τον κανονισμό. Θέλω και εγώ να τονίσω ότι ο τριμερής διάλογος ήταν ιδιαίτερα μακροσκελή. Χρειάστηκαν αρκετέ προεδρίες για να ολοκληρωθεί και τελικά εγκρίναμε τον κανονισμό επί Ρουμανική Προεδρία. Χρειάστηκε χρόνος, όπως σας είπα. Γι' αυτό θα πρέπει να επιταχύνουμε λίγο την εκτέλεση του κανονισμού αυτού. Αυτή η βασική κατεξοδότηση πράξη είναι νομικώς δεσμευτική. Και είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρακολουθεί ε, την υλοποίησή της. Άρα είναι ζωτική σημασία να δούμε τις τεχνικές πτυχές. Τι χρειαζόμαστε όταν συλλέγουμε δεδομένα. Χρειαζόμαστε υψηλής ποιότητας δεδομένα κατά πρώτον, έπειτα να είναι επίκαιρα να μην εργαζόμαστε με βάση δεδομένα που έχουν παλιώσει, μπαγιάτικα, να είναι λοιπόν επίκαιρα και μετά να έχουμε κατά απαραίτητα τεχνολογικά μέσα για να μπορούμε να τα ε, συγκεντρώσουμε σωστά. Και τα δεδομένα πρέπει να είναι και συγκρίσιμα για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας ως πολιτική όπως πρέπει. Θα στηρίξουμε λοιπόν αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κόζα. Και τώρα ο κ. Ραζέλα από τους σοσιαλιστές. Ε, ε, ευχαριστώ, ευχαριστούμε ε, εκ μέρους της κυρίας Γκρέλ να πω ότι υπάρχει μια ερώτηση για τις μελλοντικές μελέτες. θέλαμε να ξέρουμε τι θα γίνει και επίσης σε καιρούς COVID θέλαμε να καταλάβουμε τι θα γίνει με το στατιστικό υλικό Θέλουμε να δούμε αν τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν ε, να έχουμε στοιχεία προγοδότες, στατιστικά στοιχεία σε... και τι γίνεται με την τηλεργασία αυτόν τον καιρό και τα στατιστικά στοιχεία περί εργασίας. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ρινιού θέλει κάποιο το λόγο, γιατί δεν έχω κανένα στον κατάλογό μου. Από την ID Επίση όχι. Η κυρία Σντάνοκα επίση, εκ μέρου των ε, Πρασίνων. Ευχαριστώ, ελπίζω να με ακούτε. Ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση, κύριε Μέρση. Έχω αρκετές ερωτήσεις. Ιδίω για την ε, τωρινή κατάσταση, την κρίση που δείχνει και το Ευρωβαρόμετρο και το τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας ε, σε σχέση με όσα συμβαίνουν, την τηλεεργασία. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια νέα στοιχεία που περιλαμβάνει η πρότασή σα έχουν να κάνουν με τις νέες αυτές μορφές απασχόλησης, με αυτή τη νέα κατάσταση που έχει δημορφωθεί και ιδίω για τους ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες, με αναπηρίε. Και μετά μια γενικότερη ερώτηση. Μιλάμε για μοντέλα και δείκτες, ιδίως για αυτήν την περίοδο της τετραετίας. Θα μπορούσαμε να προβλέψουμε κάποιους δείκτες υποχρεωτικούς, εξειδικευμένους για μειονότητες όπως γλωσσικές μειονότητες. Η χρήση της γλώσσας εντό τη οικογένειας θα μπορούσε να είναι ένα δείκτη. Ή θα μπορούσαμε να μετρήσουμε με δείκτες τις μορφές διακριτικής μεταχείρισης με κριτήριο τη γλώσσα. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι δείκτες, αλλά όχι απευθείας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σα. Ευχαριστούμε κυρία Σντάνοκα και τώρα η κυρία Ραφάλσκα από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Πολύ κατατοπιστική. Ε, και με πολλές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των κανονισμών. Είναι σημαντικό για όλους μας και για τους ευρωβουλευτές αλλά και για τους πολίτες, διότι χρειαζόμαστε επίκαιρα στατιστικά δεδομένα που να περιγράφουν ε, κατά λεπτός τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, την πραγματικότητα που μας περιβάλλει σε καθημερινό επίπεδο. Επίσης, Χρειάζονται δεδομένα και για την ε, κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την πανδημία COVID. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι διαβουλεύσεις που μας αναμένουν ε, υπάρχει περίπτωση να είναι ιδιαίτερα μακροσκελής. Τα στατιστικά δεδομένα αφορούν την αγορά εργασίας και τις συντάξεις. φρονώ ότι οι διαβουλεύσεις θα οργανωθούν ε, στο σωστό χρονικό πλαίσιο, διότι δηλαδή δεν μας απασχολούν απλώς οι τεχνικές λεπτομέρειες. δημιουργούμε προποθέσει για τη συλλογή πολύ εξειδικευμένων πληροφοριών θα μα βοηθήσουν στο να χαράξουμε σωστά και να σχεδιάσουμε πολιτικέ και κανονισμού. Για τα ποσοστά, 5% για κάθε μεταβλητή σε οποιοδήποτε τίτλο. Αυτό ακούμε για την ώρα. Αυτό το 5% είναι αρκετό για να έχουμε τις σημαντικότερες μεταβλητές που καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες μας είναι ε, ένα σωστό όριο, σωστός περιορισμός γιατί κάποιες φορές μπορούμε να παραλύσουμε τη δουλειά των ε, θεσμικών οργάνων που συλλέγουν δεδομένα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ραφάλσκα, κάποιος εκ μέρους της ΓΚΟΕ που βρίσκεται στην αίθουσα ή θέλει το λόγο εξ αποστάσεως, remote. Κανείς. Ωραία. Να δώσω λοιπόν το λόγο και πάλι στον κύριο Μερσή ή σε μία από τις συναδέλφους του. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μέρση για να απαντήσει τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Παρακαλώ. Oui. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε. Συγγνώμη, άρχισα να μιλάω γαλλικά. γιατί ακούω τη μετάφραση στα γαλλικά. Λοιπόν, δεν κατάλαβα πολύ καλά τα όσα είπε ο κύριος Κώσα διότι είχα ένα πρόβλημα με τη διερμηνία δεν άκουγα καλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, μεγάλη σας υποστήριξη Δυστυχώς ε, έχει διακοπεί η σύνδεση του ομιλητή. Sorry, Mr. Mercy, we have... Συγγνώμη κύριε Μέρση, έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσης. Mr. Mercy, could you please press the speak button? still with... Κύριε Μέρση, παρακαλούμε, πατήστε το κουμπί speak. Δεν ακούγεται καθόλου το... η φωνή σας. So maybe we can... Λοιπόν, ενδεχομένω θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε την κυρία Γκρέλ. Κυρία Γκρέλ, αν είστε συνδεδεμένοι, θα μπορούσατε παρακαλούμε να προσπαθήσετε να μιλήσετε εσεί στη θέση του κ. Μέση, ο οποίο αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα. Ναι, είμαι συνδεδεμένη. Αλλά και εγώ είχα προβλήματα με τη μετάφραση. Δεν άκουσα την πρώτη ε, ερώτηση καλά, το πρώτο παρεμβαίνοντα. Όσον αφορά το ερώτημα του τι κάνουν οι εργοδότες για την κατοίκον εργασία, για την τηλεργασία, ήθελα να πω ότι υπάρχει μια άλλη έρευνα που συλλέγει δεδομένα για τη χρήση ε, των ε, τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών σε επιχειρήσεις. Και έχουμε και κάποιες ερωτήσεις ε, στο 20, στο 20 για τις ψηφιακές συσκευές που παρέχουν εργοδότες σε εργαζομένους και εκεί εξετάζουμε αυτό το home office τα μέσα που παρέχονται για την εργασία κατοίκων, όπως αναφέρθηκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει φτιάξει καθόλου κατάσταση με τον κύριο Μέρση. Όχι. Εξαφανίστηκε τελείως. Τον χάσαμε. Ε, Δυστυχώ θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη, αλλά πριν από αυτό θα σας ανακοινώσω την προθεσμία της ΕΜΠΛ για ενστάσεις για αυτά τα δύο θέματα. Είναι 10 Σεπτεμβρίου. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που είναι το σχέδιο γνωμοδότησης για την ανατροπή των δημογραφικών εξελίξεων στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση των μέσων της πολιτικής για τη συνοχή συντάκτρια της ΕΜΠΛ είναι η κυρία Ραφάλσκα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ραφάλσκα που δέχθηκε να εξετάσουμε στο πρωινό κομμάτι της συνεδρίας αυτό το θέμα και δίνω ακριβώς το λόγο τώρα στην κυρία Ραφάλσκα για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης για περίπου 5 λεπτά. Κυρία Ραφάλσκα, έχετε το λόγο. Ε, Κυρία Πρόεδρε, ε, κυρίε και κύριοι, το δημογραφικό αρχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα το έχει αντιληφθεί όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και άλλη και απόδειξη είναι η κατάσταση που βλέπουμε ε, για πρώτη φορά έχουμε επίτροπο αρμόδιο για το δημογραφικό. Πρόσφατα σε μια συνάντηση της Επιτροπής ε, παρουσιάστηκαν πληροφορίες για το πώς επηρεάζει το δημογραφικό θέμα άλλους τομείς της ε, ζωής. Οι δημογραφικές αλλαγές δεν σημαίνει ότι έγιναν ξαφνικά. Συντελούνται εδώ και δεκαετίες ανησυχούν τους επιστήμονες, τους οικονομολόγους, τους ε, πολιτικούς, ε, τους ειδικού σε κοινωνικά θέματα, διότι έχουν κάποιες συνέπειες, οι οποίες ε, γίνονται ήδη αισθητέ. Οι κοινωνίες στην Ευρώπη γυράσκουν. Η ηλικία είναι σήμερα 44, ενώ στο 1950, γιατί αυτή είναι η χρονική προοπτική που εξετάζουμε, ε, συγγνώμη, το 2050 θα είναι 49. Σήμερα έχουμε 20% των ανθρώπων άνω των 65 και το 2070 αυτό το ποσοστό θα έρχεται στο 30%. Και φυσικά η κατάσταση είναι διαφορετική ανάλογα με την περιοχή ή τη χώρα. Τι συνέπειες έχει αυτό. Οι δαπάνες οι οποίες ε, σχετίζονται με τις πολιτικές που σχετίζονται με τους ηλικιωμένους ε, αυξάνονται σε σχέση με τον ε, παραγωγικό πληθυσμό ο οποίος ε, σιγά σιγά λιγοστεύει σε σχέση με τους άνω των 50. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε στην γνωμοδότησή μας να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για παράδειγμα ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια από αυτά τα ταμεία για να μπορέσουν να προσαρμόσουν τον κοινωνικό κλάδο στις ανάγκες των κοινωνικών αυτών ομάδων οι οποίες αυξάνονται σε αριθμό και έχουν μεγάλες προσδοκίες. Τώρα αναφέρομαι στους ηλικιωμένου, σε οικογένειε με παιδιά. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πολύ σωστά εξετάζει ξανά το θέμα της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδολίων για την αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων ε, που προκαλεί η δημογραφική μεταβολή. Η δημογραφική αυτή μεταβολή επίσης σχεδίζεται με την ερήμωση ορισμένων περιοχών βελτιώνοντας ε, τις υποδομές μεταφορών η βελτίωση συγγνώμη, των υποδομών μεταφορών ε, και των υποδομών τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις περιοχές ε, που έχουν περισσότερους ηλικιωμένους ή που είναι πιο αγροτικές. Η πανδημία μας ανέδειξε όλα τα προβλήματα του ψηφιακού αποκλεισμού, κυρίως των ηλικιωμένων. Πρέπει λοιπόν πάση θυσία να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και αναφέρομαι τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε αυτό το ψηφιακό χάσμα των ηλικιωμένων, των πληθυσμών στις αγροτικές περιοχές. Να περιορίσουμε αυτό το χάσμα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι χρησιμοποιούμε τις ε, τεχνολογίες ε, πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών. Ε, ακόμη και εμείς που χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και τι γνωρίζουμε καλά, παρόλα αυτά μπορεί να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Ωστόσο, η πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα και διαδίκτυα δεν είναι πάντα δυνατή παντού. Ε, στο πλαίσιο λοιπόν της παιδείας, της ε, τεχνητής νοημοσύνης, ε, των δεξιοτήτων σε τεχνολογίες πληροφορικής, σε, σε όλα αυτά τα εγχειρήματα, η έλλειψη ευρυζωνικού δικτύου αποτελεί πρόβλημα γιατί σημαίνει ότι ένα κομμάτι του πληθυσμού σε κάποιες περιοχές ή σε κάποιες ηλικιακέ ομάδες εξαιρείται αποκλεί, κόπτεται από αυτές τις εξελίξεις. Θα πρέπει επίσης να κινητοποιήσουμε περισσότερα κονδύλια για να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, υπηρεσίες φροντίδας, σε αυτές αναφέρομαι τώρα. Αυτό απαιτείται λόγω της γυρένσης του πληθυσμού. Αποτελεί πρόβλημα σήμερα. Υπάρχει χάσμα μεταξύ ιδιωτικών και κρατικών υπηρεσιών φροντίδας. Αυτό σχετίζεται και με τους ανθρώπους που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα ή φροντίδα ε, όλη την ημέρα και οι άνθρωποι που υποφέρουν από μακροχρόνιες ασθένειες ε, η τηλεφροντίδα όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις χώρες που έχουν να υλοποιήσουν ορισμένα προγράμματα. Η Πολωνία αποτελεί εδώ παράδειγμα. Έχουμε το πρόγραμμα προσβασιμότητα ΣΥΝ, έτσι το ονομάζουμε, που θέλει να βελτιώσει την πρόσβαση των ηλικιωμένων ή των οικογενειών με παιδιά σε διάφορες υπηρεσίες. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά και ελπίζω η τελική έκθεση να γίνει δεκτή από εσάς. ήθελα να ζητήσω έτσι, την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ τον κύριο Φάσκα για την παρουσίαση του κειμένου, του σχεδίου. Έχουμε τώρα κάποιους και όσους που είναι συνδεδεμένοι από απόσταση είτε βρίσκονται εδώ. Από το ΕΛΚ ο κύριος Λέναρ Πίρς έχει το λόγο παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Δυστυχώς ε, ο κύριος Μάντερς είναι ο πιο της κανονικά για το ΕΛΚ. Δεν είναι εδώ όμως και μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Ραφάλσκα για αυτή την έκθεση. Κανονικά δεν προλέπονται Ολλανδικά στη συνεδρίαση αυτή όμως. Οπότε δεν μπορεί να μεταφραστούν. Πρέπει να ζητηθεί από τον ομιλητή να μιλήσει αγγλικά. Zoals ouderen. Alleen wanneer we het voorzieningenniveau op het platteland verbeteren, voorkomen we dat ouderen eh, versterkt van het platteland naar de stad trekken, waardoor Βεβαίως αν βελτιωθεί η κατάσταση στην επαρχία, οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση, καλύτερη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν να επιτρέψουν στους ηλικιωμένους να μείνουν στην χώρα τους όσο γίνεται ε, στο σπίτι του γίνεται περισσότερο καιρό, σε ένα γνωστό περιβάλλον. Έτσι πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Επιτρέπουμε στους ηλικιωμένους να νιώσουν καλύτερα ε, στο σπίτι τους και μειώνουμε και την πίεση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Στον όνομα του κυρίου Μάντες θέλω να κάνω μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει μια ανταλλαγή των πρακτικών και να ε, εντατικοποιηθεί αυτή η ανταλλαγή. Κάποια κράτη-μέλη είναι ήδη στην πρώτη γραμμή. Και όταν κάποιες πρακτικές καινοτόμες ε, ε, βοηθούν την κατάσταση, ε, θα πρέπει να, με, να όλοι μας και πρέπει βεβαίως τα άτομα, τα ηλικιωμένα να συμμετέχουν περισσότερο στην, στα κοινά και στον πολιτικό κόσμο, αν θέλεις, διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που γνωρίζουν τι χρειάζονται καλύτερα. Ε, ο κ. μάντερ χαίρεται που υπάρχει και το κοινοβούλιο των ηλικιωμένων. Πρέπει λοιπόν οι ηλικιωμένοι να, να ακουστεί η φωνή τους. Υπάρχει το κοινοβούλιο των νέων. Ένα κοινοβούλιο των ηλικιωμένων ε, θα ήταν μια καλή ιδέα, διότι θα επέτρεπε για άλλη μια φορά ανταλλαγή βάση των πρακτικών για να μπορέσει κάποιο να γεράσει με υγεία ε, να παραμείνουν δυνατότητε για του ανθρώπου αυτού, να υπάρχουν δυνατότητε και στην ύπεθρο Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του κόστου και επίση θα μπορέσουν οι ηλικιωμένοι να μεταδώσουν τι γνώσει του στου πιο νέου. Ε, η κυρία Ραφάλσκα και ο κ. Μάντε ε, θα είναι καλό να συνεχίσουν να συνεργάζονται για το ζήτημα αυτό. Από το S&D ο κ. Μπέργκερ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε αυτό το σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική έκθεση. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια που γίνεται αντιμετώπιση αντιμετώπισης των δημογραφικών αλλαγών. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις. Υπάρχει ένα ψήφισμα ήδη από το 2011 για τις δημογραφικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους για, τις μελλοντική, για πολιτική συνοχής και υπάρχει και ένα άλλο ψήφισμα του 2017 για την χρήση των ε, εργαλείων κοινωνικής πολιτικής ως απάντηση στη δημογραφική αλλαγή. Νομίζω πως είναι σημαντικό να πιέζουμε διαρκώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους ιδιαίτερα τα μέσα πολιτικής συνοχής για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτήν τη δημογραφική τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει και σε μια μείωση ε, του χάσματος που υπάρχει στην εξέλιξη από τη μια χώρα στην άλλη το, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή διότι κάποιες περιοχές, κάποιες περιφέρειες αυτή τη στιγμή ερημώνουν και εκεί υπάρχει και έλλειψη πολύ βασικών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη της πανδημίας ε, αποκάλυψε Αυτέ τις ελλείψει, αυτά τα προβλήματα με τρόπο εξαιρετικά επώδυνο. επώδυνο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες ε, και, και έχουμε το κίνητρο για να το κάνουμε αυτό, διότι είδαμε τι συμβαίνει στον κόσμο όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στι δημόσιες υπηρεσίες για όλους, ιδιαίτερα για όσους ε, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη των υπηρεσιών, τα παιδιά, όσοι ε, πλήττονται ε, ή ε, έχουν κάποια χρόνια ασθένεια, οι πιο ηλικιωμένοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτές τις βασικές υπηρεσίες που να είναι προσβάσιμες σε όλους. Επίσης η πανδημία μας έδειξε ότι ε, μπορεί να δημιουργηθεί πολύ μεγάλη ζημιά ε, και για τους ανθρώπους που περιθάλπτουν τους ηλικιωμένου άτυποι νοσηλευτέ στα σπίτια τους. Θα πρέπει να επαναλάβω ότι η δημογραφική αλλαγή θα πρέπει να αποτελεί μέρος ε, όλων των προτεραιοτήτων μας. Ε, κοινωνική αλλαγή, ε, κοινωνική Ευρώπη, έξυπνη Ευρώπη, πράσινη Ευρώπη, όλα αυτά σχετίζονται με τις δημογραφικές αλλαγές. Είναι ένα οριζόντιο ζήτημα. Θα προσπαθήσω λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία να τα συμπεριλάβω στην έκθεση, θα συνεργαστώ στενά μαζί σας, θα πρέπει να έχουμε μια ισχυρή έκθεση που θα βασίζεται στα δικαιώματα. Ευχαριστώ για το Renew τώρα. Ο κύριος Κάνιας έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία Ραφάλσκα για το έργο της. Πρόκειται για μια έκθεση με έναν τίτλο πολύ σημαντικό. Να επενδύσουμε, μάλλον να αντιστρέψουμε τις δημογραφικές ε, περιοχές χρησιμοποιώ, ε, τις δημογραφικές, αλλά, δημογραφικές τάσεις ε, χρησιμοποιώντας ε, τις, ε, τα εργαλεία κοινωνικής συνοχής. Είναι δύσκολο βεβαίως να έχουμε άποψη πάνω σε μια έκθεση που δεν υπάρχει ακόμα. Θα ήταν καλό να έχουμε την έκθεση για να μπορέσουμε να κάνουμε συστάσεις που να έχουν να κάνουν ε, νόημα. Και αυτή την έκθεση από ό,τι φαίνεται δεν θα την έχουμε έως τις αρχές Οκτώβρη. Το λέω αυτό για να πω ότι οι προτάσεις που κάνουμε εμείς τώρα στην ομοδότηση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, δεν βασίζονται μάλλον σε κάποιο έγγραφο. Η γνωμοδότηση θα πρέπει να βασίζεται σε μια έκθεση την οποία δεν έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Ε, το θέμα της γύρανσης της Ευρώπης είναι μια από τις προκλήσεις για την Ευρώπη. Ε, και ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες όπου αυτή η γύρανση συνδέεται με την, με την ερήμωση. Χαν φεύγουν νέοι άνθρωποι, ε, εκεί, οπότε ο μέσος όρος ανεβαίνει ε, των ε, κατοίκων και επίσης μειώνεται οι κάτοικοι. πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν στις περιοχές εκείνες όπου αυτή η τάση γύρανσης οδηγεί και σε ερήμωση. Και εδώ έχουμε ένα νέο πρόβλημα. Έχουμε αφενός ε, τη γύρανση και αφετέρου την, τον αφανισμό χωριών ολόκληρων, περιοχών, δήμων. Σε εθνικό επίπεδο ε, υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ένα χρέος απέναντι σε αυτές τις περιοχές. Τις έχουμε εγκαταλείψει συστηματικά σε πολιτικό επίπεδο και αυτό το χρέο θα πρέπει κάποια στιγμή να το αποπληρώσουμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι περιοχέ εκείνε που χρειάζονται επενδύσει. Χρειάζεται ένα κατάλληλο επίπεδο επενδύσεων όχι μόνο για να σταματήσει η τάση αυτή αλλά να αντιστραφεί. Στην Ισπανία υπάρχουν πάνω από χίλια, χίλιοι δήμοι χωρίς παιδιά κάτω 4 ετών. Ε, πολλές, πολλοί δήμοι με λιγότερο από 20 κατοίκους, χωριά που εξαφανίζονται. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό στην έκθεσή μας, είναι στην επιτροπή μας είναι σημαντικό αυτό που θα προτείνουμε, διότι μόνο αν μπορέσουμε να δώσουμε ευκαιρίες, δυνατότητες στις περιοχές αυτές, θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε την τάση αυτήν. Απασχόληση λοιπόν και κοινωνικές υπηρεσίες. Απασχόληση σε ψηφιακό τομέα, τηλεαπασχόληση, ε, αυτά μπορούν να βοηθήσουν στο να αλλάξουν πολύ τα πράγματα. Και αυτό αυτέ είναι οι βασικέ στρατηγικέ γραμμέ τη επιτροπή μα και αυτού του Κοινοβουλίου. Η ψηφιακή Ευρώπη και πράσινη Ευρώπη. Εάν μπορέσουμε να βελτιώσουμε τι επενδύσει συγκεκριμένες πολιτικές πολιτικέ της απασχόληση, βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, των υγειονομικών υπηρεσιών ε, και των υπηρεσιών περίθαλψη, μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση και να έχουμε μια Ευρώπη πιο δίκαια και πιο ολοκληρωμένη και πιο ισορροπημένη. Uh, on behalf of... Και τώρα, εκ μέρους της ID, η κυρία Μπίλντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, εισηγητή. Δυστυχώς έχουμε ξαφνικά πολύ κακό ήχο στη σύνδεση. Yes, we do have some technical... Έχουμε τεχνικό πρόβλημα με τη σύνδεσή σας, κυρία Μπίλ, τη λέει η Πρόεδρος. Ίσως αν χρησιμοποιούσατε ακουστικά, διότι είστε σε μεγάλη αίθουσα. Και τώρα πάλι δεν με ακούτε. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, αλλά με πολύ κακό ήχο, δυστυχώς. There is a lot of background noise. You would have to... You would have to... Δυστυχώς υπάρχει ηχό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλα ακουστικά. Well, for now we will switch, Madam Bilde. We'll get back to her and... Δεν μπορούμε για την ώρα να ακούσουμε την κυρία Μπίλ. Θα την ακούσουμε αργότερα και τώρα κυρία Σντάνοκα. Με ακούτε. Για μας τους πρασίνους Όταν μιλάμε για την ελληνική μεταξύ των γενεών και την γύρευση του πληθυσμού, τα στατιστικά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Οι ηλικιωμένοι, οι μονογονέικες οικογένειες, οι άνθρωποι με αναπηρίες, οι φτωχές οικογένειες, τα νοικοκυριά σε συνθήκες ένδυας, είναι οι ευπαθείς ομάδες που αφορούν ιδιαίτερα τα στατιστικά αυτά στοιχεία για τις πολιτικές συνοχής. Γιατί αυτού στοχεύουμε. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και συγκεκριμένοι δείκτες για τις γυναίκες ας πούμε, στατιστικά στοιχεία για τις δημογραφικές αλλαγές και όπως είπαν ήδη πολλοί συνάδελφοι, υπάρχουν ε, περιφερειακές πτυχές για περισσότερο ή λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής Υπάρχουν περιφέρειες που πρέπει να λάβουν ε, αυξημένη προσοχή. Σε ό,τι αφορά κάποια θέματα που έθιξαν οι συνάδελφοι από τους ισοελιστές και δημοκράτες για την ε, αλλαγή στις δημογραφικές τάσεις και το τι θα πρέπει να κάνουμε ε, το reversing, δηλαδή η ε, αντιστροφή των δημογραφικών τάσεων, δεν είναι σωστή πολιτική. Η δική μας η πρόταση είναι να έχουμε μια πιο θετική αποτίμηση και προσέγγιση. Να δημιουργήσουμε δηλαδή τέτοιες προϋποθέσεις που να στηριχθούν οικογένειες που να επιτρέψει στις οικογένειες λοιπόν που υποστηρίζονται να αποφασίσουν μόνες τους τι οικογενειακό σχεδιασμό θέλουν, πόσα παιδιά θα έχουν, πώς θα ζήσουν τη ζωή τους, τι σχέδια θα έχουν για το μέλλον και πώς θα είναι η οικογένειά τους. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ραφάλσκα για την παρουσίασή της, για τις προτάσεις της την ακούσαμε Δεν είναι ακόμα περατωμένη η έκθεση, αλλά μαζί πιστεύω μπορούμε να συνεργαστούμε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε κυρία Σντάνοκα. Με την κυρία Build. Πώς πάει η σύνδεση. Ας ξαναπροσπαθήσουμε. Κυρία Build, έχετε το λόγο. Μ' ακούτε. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Η Ευρώπη ε, αρχίζει να χάνει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού πληθυσμού της. Και είναι ένα γεγονός. Ε, γιατί, γιατί έχουμε λιγότερα παιδιά. 1,6 είναι το ποσοστό γονιμότητας, ο συντελεστής γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευθύνει διαρκώς. Η Γαλλία είναι στο 1,89% πρώτη των πρώτων στην Ευρώπη, αλλά δεν αρκεί αυτό για την ανανέωση του πληθυσμού στην Ήπειρο. Πολλές είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν ποσοστά τα οποία είναι σε δραματική πτώση και μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι θα ανεγείρονται σοβαρέ ανησυχίε για τι επόμενε δεκαετίε. Έχουμε περισσότερου θανάτου από ό,τι γεννήσει το 2020. Και όμω ο πληθυσμό δεν πάβει να διωγγώνεται. Ο λόγο είναι απλό, οι μετανάστε. Εδώ βρισκόμαστε στην καρδιά του θέματο, ενώ οι προτάσει που γίνονται στα πλαίσια του κειμένου αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψουν ε, στα ε, δημογραφικά να επηρεαστούν ε, σε όλε τι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετανάστευση θα έχει μια ιδιαίτερη μεταχείριση μετανάστευση. Ε, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα δύο, τις δημογραφικές τάσεις από τη μετανάστευση. Πρέπει λοιπόν να μην παρουσιάζουμε τα πράγματα διαφορετικά, ε, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση. Οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας είναι οι εξή. Είτε δεχόμαστε να είμαστε λιγότερο πολυάριθμοι και να διοργανωθούμε διαφορετικά, προστατεύοντας όμως την ταυτότητά μας, είτε αποφασίζουμε να ε, επιτρέψουμε την είσοδο εκατομμυρίων μεταναστών, δημιουργώντας όμως αμετάκλητες και βαθιές αλλαγές στις κοινωνίες μας. Εμείς αρνούμαστε αυτό το μονόδρομο. Υπάρχουν και άλλε επιλογέ. Οι πολιτικοί συνοχή δεν θα λύσουν μόνο του το πρόβλημα. Τα δημογραφικά δεν μπορούν να βρίσκονται μόνο στην καρδιά τη δράση μα ε, χωρί να έχουμε αυτέ τι φιλοδοξίε. Η δική μα ε, ομάδα, ε, το, το δικό μα κόμμα, το Rassemblement Νασιονάλ και η συμμαχή μα, θέλουμε να έχουμε φιλοδοξότερου στόχου. Όχι απλώ το στενό πλαίσιο όσων εδώ περιλαμβάνονται. Η Ευρώπη των αξιών των αρχών της κληρονομιάς μας είναι η Ευρώπη της ιστορίας μας που θέλουμε να προστατεύσουμε. Γιατί να κοιτάμε τι θα γίνει στο μέλλον αν έχουμε ήδη απαρνηθεί την ίδια μας την ύπαρξη συλλογικώς. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Από την ΚΟΥ έχουμε τον κύριο Μποτέγκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την κυρία Ραφάλσκα, την ε, εισηγήτρια. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει σημαντική κινητικότητα μεταξύ ε, επαρχίας και πόλεων ε, και μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών την τελευταία δεκαετία μου είπαν ότι πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από την ανατολική πλευρά της Υπήρου προς τη δυτική και δεν είναι από ελεύθερη επιλογή. Όταν στην Κροατία υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία στα γερμανικά δεν είναι γιατί όλοι αγαπούν τα γερμανικά. Όταν οι Ιταλοί του Νότου θέλουν να έρθουν στις Βρυξέλλες δεν είναι μόνο διότι τους αρέσει το κλίμα στις Βρυξέλλες, αντιθέτω είναι γιατί δεν βλέπουν να έχουν μέλλον εκεί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχουν καλές κρατικές υπηρεσίες, καλές θέσεις εργασίας, πολύ χαμηλή μισθή, ε, δεν τους επιτρέπουν να ζήσουν. Οπότε η απάντηση της Κομισιόν είναι διαρθρωμένη, την είδαμε ε, την περασμένη εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είπε ρητά ότι προτείνει δύο μεγάλες πολιτικές επιλογές. Η πρώτη είναι το να φέρει το διαδίκτυο σε περιοχές που ερημώνονται αυτή την εποχή πολύ καλά, αλλά είναι σαφές ότι αυτό δεν αποτελεί απάντηση ε, σε θέματα κρατικών υπηρεσιών και απασχόλησης και μετά ε, η αγορά, η οικονομία των ε, υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Μαζική επένδυση στις κρατικές υπηρεσίες, συγκοινωνίες, ταχυδρομεία σε χωριά, συντάξεις κτλ. Και δεύτερον φυσικά θέσεις απασχόλησης ποιότητας σε όλη την Ευρώπη. Και εκεί πιστεύω ότι απαιτείται μια βιομηχανική πολιτική πολύ περισσότερο από τα ταμεία συνοχής, η οποία θα εγγυάται αυτή η βιομηχανική πολιτική την εργασία και θα την κατανέμει με τρόπο ισότιμο στην ευρωπαϊκή επικράτεια, αντί να την επικεντρώνει σε ορισμένους πόλους ανταγωνιστικότητας, όπως ονομάζονται τώρα. Αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και ε, με γνώμονα αυτό θα συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή την έκθεση και ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπότσκορ από το ΕΛΚ ήθελε να πάρει το λόγο. Ε, κυρία Μπότσκορ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Can you hear me now? Hello? Yes. Με ακούτε τώρα, ναι, σας ακούμε. Uh, thank you very much for... Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Θα ήθελα να σχολιάσω εν συντομία αυτό το θέμα και θα μιλήσω ουγγρικά αφού υπάρχει μετάφραση. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ραφάλσκα για την γνωμοδότηση αυτή και πρέπει να πω ότι Συμφωνώ με όλους όσοι μίλησαν και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουμε να ανατρέψουμε τις δημογραφικές τάσεις στην Ευρώπη διότι φοβάμαι ότι μέχρι το 2070 ο πληθυσμός της Ευρώπης θα έχει πέσει σε λιγότερο από 4% του παγκοσμίου πληθυσμού. Είναι σοκαριστικός ο αριθμός αυτός. Η Ευρώπη γυράσκει όπως γνωρίζουμε όλοι και ναι θα πρέπει να προσέχουμε τα ε, νούμερα αυτά. Συμφωνώ επίση με όσους είπαν ότι χρειάζεται να επενδύσουμε, να δημιουργήσουμε θέσει εργασία. και ότι χρειάζεται να ε, πάμε τις ε, υπηρεσίες, τις κοινωνικές υπηρεσίες σε περιοχές που γυράσκουν και να προσελκύσουμε τις νέες γενιές στις περιοχές αυτές. Αλλά είναι πολύ σημαντικό όχι απλά να ενθαρρύνουμε την κίνηση των ανθρώπων προς αυτές τις περιοχές, τις αγροτικές περιοχές, αλλά να επιμείνουμε και στη δημιουργία οικογένεια μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να του βοηθήσουμε δηλαδή να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένειε. Πρέπει να, δείξουμε, να δείξουμε ε, τι θετικέ πτυχέ τη ε, οικογενειακή ζωή. Την τελευταία δεκαετία η εικόνα αυτή έχει υποβαθμιστεί διότι η ατομικότητα πλέον έχει προτεραιότητα και το μοντέλο της οικογένειας έχει μείνει στο παρασκήνιο, ειδικότερα στις μεγαλοπόλεις. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το οικογενειακό μοντέλο και να το προωθούμε. Να βοηθάμε οικογένειες ε, με κάποιες ε, ε, υπηρεσίες, με κάποια οικονομική βοήθεια, με βοήθεια για να αγοράζουν σπίτι, υποστήριξη για την δημιουργία οικογένειας ή να τους βοηθάμε να μπορούν να συνεχίσουν τα παιδιά τις σπουδέ. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να εξαναγκάσει κανέναν να κάνει μεγάλη οικογένεια ή να αποκτήσει παιδιά. Αλλά πιστεύω ότι αν φτιάξουμε το σωστό οικονομικό υπόβαθρο για κάτι τέτοιο, τότε οι νέοι άνθρωποι είναι περισσότερο να έχουν μια καλή ευκαιρία να δημιουργήσουν μια οικογένεια. Ευχαριστούμε κύριε Μπότσκον. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της DG Regio από την Κομισιόν που πρέπει να έχει συνδεθεί. Please press the speak button. Παρακαλώ πατήστε το κουμπί ομιλίας. Ο κύριος ε, Κυμπορόπουλος, παρακαλώ. Συγγνώμη, όχι, Τέριστερόπουλος από την DG Radio. Δεν είναι ο κύριος Κυμπορόπουλος, έκανα λάθος ομιλήτρια. No connection. Okay, never mind. Δεν υπάρχει σύνδεση, δεν μπορούμε. Λοιπόν, για να κλείσουμε, δίνουμε το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ραφάλσκα, παρακαλώ. E, dzięki mm, temu, że nie możemy się połączyć zdalnie, będę miała więcej. Δεν έχουμε καλή σύνδεση. Οπότε αυτό μου δίνει περισσότερο χρόνο για να δώσω απαντήσει σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ για όλα τα επιχειρημάτα που ακούσαμε. Μερικές φορές ε, απέχουν αρκετά το ένα από το άλλο γεγονός που δείχνει ότι το θέμα ε, το δημογραφικό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και θα πρέπει να βρούμε κάπου κάποια μέση λύση. Φυσικά είναι δύσκολο να εκδώσει κανείς μια γνωμοδότηση όταν δεν είναι ακόμα έτοιμη η έκθεση. Ε, αλλά έχουμε δημογραφικά δεδομένα για διάφορες ε, χώρες ή μέσους όρους ε, ε, για ολόκληρη την Ευρώπη. Ρωτήθηκε κάτι βασικό, πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε τις τάσεις και αν αυτό είναι δυνατόν. τι μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτή την αργυρή οικονομία, την γκρίζα οικονομία να μην γίνει, να μην γίνει ακόμη πιο γκρίζα. Το ποσοστό γενετικότητας είναι πολύ χαμηλό. Στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα δεν θα καταφέρουμε να ανανεώσουμε τις γενιές γιατί βρίσκεται γύρω στο 1 ενώ χρειάζεται να είναι 2,1 ο δείκτης αυτός. Φυσικά οι κοινωνικές πολιτικές είναι αρμοδιότητες των κρατών μελών. Ωστόσο, μπορούμε να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες ε, για τη δημιουργία οικογένειας. Όταν κάποιος θέλει να αποκτήσει παιδιά, θα πρέπει να του προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες. Αυτό σχετίζεται με τις κοινωνικές πολιτικές λοιπόν, με την ε, πολιτική της αγοράς εργασίας ή της στέγασης. Ε. Σίγουρα δεν πρέπει να ξεχνάμε κανέναν από αυτούς τους τομείς. Έχουμε την καταστρεπτική ε, απερίμωση ορισμένων περιοχών. Ο κόσμος φεύγει από εκεί. Κάποιοι υποφελούνται φυσικά από αυτή, τον αποπληθισμό, οπότε πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, πολιτικές ε, για αυτό το ζήτημα. Ε, ερωτήθηκε, υπόθηκε κατά πόσο ότι η πολιτική συνοχή δεν μπορεί να μας βοηθήσει να αντιστρέψουμε το δημογραφικό τις δημογραφικές τάσεις. Εγώ ουδέποτε πίστεψα ότι τα οικονομικά μέσα ή η πολιτική συνοχή είναι τα μόνα εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιστρέψουμε αυτές τις ε, τάσεις. Το μόνο που κάνουμε εδώ είναι ότι υποστηρίζουμε ε, αυτή την ε, θετική εξέλιξη. Πολλοί κόσμος αναφέρθηκε στην διαγενειακή αλληλεγγύη. Πιστεύω ότι όλα τα μέσα της Επιτροπής ΕΜΠΛΕ υποστηρίζουν την ιδέα αυτή. Ο κόσμος ζει περισσότερο. Αυτό είναι γεγονός και είναι καλό αλλά θέλουμε επίσης να βελτιώνεται και η ποιότητα ζωής. Το να παραμένει κανείς υγιής θα πρέπει να είναι δυνατόν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής κάθε ανθρώπου και εδώ έχουμε σοβαρές διχογνωμίες και σοβαρές διαφορές. Οι συνταξιούχοι στην Ανατολική, στην Κεντρική Ευρώπη ε, ακόμα ζουν υγιώς ε, για λιγότερα χρονικό διάστημα από ότι στη Σουηδία ή στη Γερμανία που τα συστήματα υγείας είναι πολύ πιο εξελιγμένα. Εδώ παρατηρήσαμε ένα πρόβλημα το οποίο ανέδειξε η πανδημία και αυτό είναι ένα από τα καλά της πανδημίας είναι ότι τι γίνεται με τον τομέα της φροντίδας, φροντίδα των παιδιών ή των ηλικιωμένων. Θέματα αρκετά σημαντικά για πολλές ε, ευρωπαϊκές χώρες. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να διατίθενται τόσο ιδιωτικά όσο και δημοσίως σε επίπεδο ποιότητας επαρκές. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή σε αυτό το κλάδο της αγοράς εργασίας και να δώσουμε και λύσεις. Τώρα, συζητάμε περί πολιτικής για τους ηλικιωμένους που αποτελεί επίσης αρμοδιότητα των κρατών μελών αλλά όλες οι δραστηριότητες οι οποίες ε, σχετίζονται με την πολιτική συνοχή, όπως η βελτίωση της πρόσβασης σε κοινωνικές υποδομές, σε υποδομές μεταφορών, σε ποιοτικά συστήματα υγείας τα οποία να είναι και ανθεκτικά σε περιπτώσεις πανδημίας ή οικονομικής κρίσης. Όλα αυτά μπορούν να ληφθούν υπόψη σε πολλούς διαφορετικούς τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήσαμε επίσης ε, περί αγοράς εργασίας διότι η αλλαγή της ηλικιακής δομής της κοινωνίας έχει ως αποτέλεσμα στην έλλειψη ε, εργατικών χεριών σε ορισμένες περιοχές. Η εργατικού δυναμικού γενικότερα. Επίσης έχουμε τη μετανάστευση των νέων και σε κάποια μέρη βλέπουμε ότι σε εποχές πανδημίας οι απασχολούμενοι μεγαλύτερης ηλικία ε, κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους. Εάν δεν αντιστρέψουμε τις τάσεις αυτές, τότε δεν θα καταφέρουμε, θα πρέπει να μετριάσουμε κάπως αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα αντιστρέψουμε όλες αυτές τις στάσεις Στο μέλλον ε, προσαρμοσμένα στις δομές της κάθε χώρας και περιοχής φυσικά. Όλα αυτά απαιτούν ευέλικτη στάση όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές και ε, επιδεξιότητα στην επιλογή των απαραίτητων μέσων βάσει σωστής ποιοτικής έρευνας και αξιολόγησης ε, της κατάστασης σε κάθε περιοχή. Πιστεύω ότι ο καθένας βλέπει διαφορετικά τις ε, κοινωνικές πολιτικές και ειδικότερα πρέπει να βλέπουμε διαφορετικά τις κοινωνικές πολιτικές όσον αφορά τις οικογένειες και τους ηλικιωμένους. Αλλά πιστεύω θα πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε εδώ σε αυτή την Επιτροπή έναν κοινό παρονομαστή που θα μας βοηθήσει να αντιστρέψουμε ή να μετριάσουμε αυτές τις αρνητικές τάσεις που συχνά παραβλέπουμε. Πρέπει να το παραδεχθούμε. Πάντα υπάρχουν πιο επίγοντα ζητήματα, αλλά θα πρέπει να τα δούμε σοβαρά και να βρούμε λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά όλους για τα σχόλια και την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ. 16 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία ε, η υποθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και τώρα περνάμε στο σχέδιο έκθεσης ε, για την ε, Ευρωζώνη 2020 θα σας δώσω το λόγο για να παρουσιάσετε το σχέδιο γνωμοδότησης κυρία Ντόμπρεφ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την σπουδαία δουλειά που έκαναν έως τώρα λάβαμε 406 τροπολογίες και όλες αυτές είναι εξαιρετικά περίπλοκες και σημαντικές. Νομίζω ότι θα φτάσουμε ένα συμβασμό τελικά και η έκθεση θα είναι μια δυνατή έκθεση έτσι ώστε να ε, δημιουργήσουμε από κοινού τις μελλοντικέ ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης. Θα ήθελα να πω ποια είναι τα σημεία ε, όπου πάμε προς σύγκληση και τα σημεία εκείνα όπου ακόμα θα πρέπει να γίνουν αρκετές συζητήσεις, επικοδομητικές πάντα βέβαια. Από ό,τι φαίνεται όλα τα κράτη-μέλη, συμφωνούμε όλοι, όλοι τα κράτη-μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλους τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους για να μετριάσουν την κρίση. Αλλά και να εφαρμόσουν καλύτερα τις συστάσεις αναχώρα και να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID είδαμε πόσο σημαντικό είναι οι πολιτικές μας να εστιάσουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, να ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο, ιδιαίτερα όταν έχουμε νέους ε, τρόπους ε, και συνθήκες εργασίας και να έχουμε δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλους. Νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμβασμό τελικά σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον ελάχιστο μισθό, τον κατώτατο μισθό, ένα σημαντικό ζήτημα θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων ε, για να επιτευχθούν και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξη των ΗΕ και το πράσινο, ε, το Green Deal το ευρωπαϊκό. Όλες οι τροπολογίες που είδα ε, πάνε προς αυτή την κατεύθυνση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και βεβαίως μιλούσαμε, μιλήσαμε για αυτό το θέμα τόσο καιρό που οι ψηφιακέ πτυχέ, οι πράσινε πτυχέ, οι οικονομικέ πτυχέ τη πολιτική μα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο, πρέπει να είναι η ίδια προτεραιότητα, να είναι η ίδια σημασία με την κοινωνική διάσταση των πολιτικών μα. Η, η κρίση μα έδειξε πώ οι ευάλωτε ομάδε, πώ οι άνθρωποι που έχουν λιγότερη κοινωνική προστασία βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση όταν μια κρίση όπω η κρίση του COVID, οποιαδήποτε άλλη οικονομική κρίση ή οποιαδήποτε άλλη έκτακτη κατάσταση προκύπτει. Και έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία τώρα όπου πιστεύω ότι θα είναι πιο δύσκολη η συζήτηση, επικοδομητική όμως πάντα επαναλαμβάνω. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο νομικό εργαλείο. Κατά πόσο θα είναι πλαίσιο, ομω παντα επαναλαμβανω πόσο θα είναι οδηγία ε, για το ε, κατώτατο μισθό ή για τις συνθήκες εργασίας. Πάντα αυτό το ζήτημα ε, οδηγεί σε δύσκολες συζητήσεις. Δεν κρύβω την άποψή μου ότι θεωρώ ότι οι κοινωνικές πτυχές, οι κοινωνικοί κανόνες πρέπει να είναι υποχρεωτικοί, τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπω ότι υπάρχει διαφωνία, υπάρχει απόκληση απόψεων ε, για το θέμα ε, της ε, ασφάλισης για την ανεργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρω ότι είναι προτεραιότητα της κυρίας Βοντελέιν αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Εκεί όμως που βλέπω το μεγαλύτερο αγκάθι, όχι μόνο στην Επιτροπή μας, αλλά και σε άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου, είναι το κατά πόσο, μεταρρύθμιση του, του, κατά πόσο χρειάζεται μεταρρύθμιση του Συμφώνου σταθερότητα και Ανάπτυξης ε, και του... Ε, ε οικονομικού οικοδομήματος που έχουμε. Κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει επαρκής ε, κάλυψη, υπάρχει επαρκής ευελιξία. Όμως η πλειοψηφία, μεταξύ των οποίων και εγώ, θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να μεταρρυθμιστεί το σύμφωνο σταθερότητας και χαίρομαι που έχω στα χέρια μου την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού ε, Οργανισμού που λέει ότι πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις ε, είναι απαραίτητες για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης, ιδιαίτερα οι χώρες που έχουν επηρεαστεί πιο έντονα, που χτυπηθεί περισσότερο από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν ήταν αρκετά έτοιμα, ακόμα και σε χώρες με, υψηλό με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χώρες. Αν όμως κάποιος δεν έχει ένα σταθερό, ισχυρό κοινωνικό σύστημα ασφάλισης, ένα σύστημα υγείας, ε, τότε αν δεν υπάρχει ένα δίκτυο αλληλεγγύης, ε, τότε τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το ζήτημα προ, πρωτίστως κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ και τώρα να περάσουμε στους κοιόδης ηγητές ξεκινώντας ε, με τον κύριο Κόσα ίσως. Είναι εδώ ο κύριος Ράτκε. Ο κύριος Ράτκε έχει το λόγο. Παρακαλώ. Mr. Radke, please press the speak. Κύριε Ράτκε, παρακαλώ. Mr. Ratke, your microphone is not working. Κύριε Ράτκε, δεν λειτουργεί το μικρόφωνο σας ε, για την ώρα. Αριστερά είναι το κουμπί. Okay, we'll solve this problem uh, lately now. Μάλιστα, θα λύσουμε το θέμα αυτό στη συνέχεια. Η κυρία Μπρουνέ τώρα από τη Renew. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα, με ακούτε? Κυρία Πρόεδρε, Θα μιλήσω στο όνομα του συναδέλφου από τη Renew που δεν μπορούσε δυστυχώ να συμμετάσχει σε αυτή την αλλαγή απόψεων και μου ζήτησε να σα μεταφέρω κάποια στοιχεία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την κυρία Ντάμπρεφ για το σχέδιο έκθεσης. Πολλέ τροπολογίες έχουν υποβληθεί και δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Οι συναδέλφου τη ομάδα Renew έχουν υποβάλει και εμεί τροπολογίε, έτσι ώστε ε, η απασχόληση, το κοινωνικό στοιχείο είναι προτεραιότητα. Για μας τρεις είναι προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα ε, θα επίγει να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας, να υποστηρίξουμε την απασχόληση, να, να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Το σχέδιο ανάκαμψης, το ιστορικό που εγκρίθηκε τον Ιούλιο, πρέπει να, να στηρίξει τους πιο επισφαλείς, τους πιο νέους, τους πιο, ε, τους πιο τροτούς για να διαφυλάξουμε τις συνθήκες εργασίες τους. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι να έχουμε πάντα ένα σωστό προσανατολισμό μακροπρόθεσμα. Είναι κρίσιμο οι πολιτικέ, οι οικονομικέ, οι δημοσιονομικέ, οι κοινωνικέ να οδηγούν στην επίτευξη των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη θέσπιση τη πολιτική μα ανάπτυξη, όπω προβλέπεται η πράσινη ανάπτυξη, ε, το, το Green Deal, και βεβαίω η ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τρίτη προτεραιότητα πρέπει να ενισχυθεί η εφαρμογή τη κοινωνική ατζέντα. Η κρίση ε, αποκάλυψε τι ανισότητε, ε, τι ε, αδυναμίε του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτήν την κοινωνική ατζέντα. Ω παράδειγμα, να πω ότι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο για ένα ελάχιστο μισθό, το οποίο αναφέρθηκε σε κάθε κράτο μέλο, ή ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό ασφάλιση ανεργία είναι απαραίτητα. Ε, είμαι βέβαιη ότι ήδη αύριο θα βρούμε συμβιβασμούς με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτό το σαφές μήνυμα υπέρ της κοινωνικής Ευρώπης να το μεταφέρουμε. Ε, κάτι που το οποίο χρειαζόμαστε όλοι σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Μπρινέ και τώρα να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Ράτκε. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. τον κύριο Ράτκε για την ώρα, οπότε συνεχίζουμε με την κυρία Ζαμέ από τους ID. Alors, <clears throat> Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρία εισηγήτρια, όντως οι τροπολογίε είναι κάποιες περίπλοκες γι' αυτό θα κοιτάξω να δώσω κάποιες εξηγήσεις Και για μας είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας, ιδίω των ευπαθών ομάδων από κοινωνικής ή οικονομικής Όμω, Όμως ε, στην έκθεση αυτή βλέπουμε πάλι ο φεντεραλισμός να πρετανεύει. Ε, πάλι έχουμε τα ίδια δογματικά ε, και ιδεολογικά συμπεράσματα. Βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών όμω. Η Ευρωζώνη έχει τα χαμηλότερα ποσοστά ανάπτυξη παγκοσμίω. Το συζητάμε όλο το πρωί. Είμαστε η περιοχή όπου υπάρχει περισσότερη δυσπιστία για το μέλλον. Γι' αυτό οι βουλευτές της ομάδας μας, Ταλή και ε, θελήσαμε να υποβάλουμε μια σειρά τροπολογιών για να ζητήσουμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να διευκρινιστεί το κατά πόσο η διοργάνωση της αγοράς εργασίας είναι αρμοδιότητα εθνική των κρατών μελών, συγκεκριμένα για το θέμα του ελάχιστου μισθού. Είμαστε κατά της ε, άποψης του κατώτατου μισθού, του ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού, που πολλές φορές βλέπουμε να αναφέρεται ε, ανάγλυφα εδώ στο κείμενο. Θα πρέπει ε, πολιτικές της Ευρωζώνης να κοιτάξουν την ε, πολιτική απασχόληση κατά πρώτο λόγο, κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει. Ε, μέχρι τώρα οι πολιτικές που είχαν εφαρμοστεί είχαν μεγάλο αντίκτυπο, αλλά δυστυχώς πολύ δραματικό και ε, πραγματικά ε, θα πρέπει να επιστρέψει η εξουσία και δύναμη στα χέρια του λαού, για το λαό και για το δικό του το συμφέρον. Ε, θα πρέπει εδώ λοιπόν να ξαναμπεί το συμφέρον των πολιτών στο κέντρο ε, κειμένων όπως αυτό που μας προτείνεται. Πρόεδρε, συνάδελφε, ε, συνάδελφοι, είμαστε πεπισμένοι η μόνη μας ελπίδα είναι να διατρανωθεί και πάλι η έννοια του έθνους. Είναι ο μόνος τρόπος για να διεξαγάγουμε μια πολιτική ε, οικονομική χρήσιμη και βάση της ε, αγαστής συνεργασίας μεταξύ των κρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ζαμέ. Από τους Πρασίνους έχουμε την κυρία Ζήπεν. Langen are you Κυρία Ζήπεν, είστε εκεί. Okay. Δεν την έχουμε την κυρία Langen -Zippen. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Γκόικινγκ, αν και δεν είμαι σίγουρος την εδώ, ούτε εκείνο είναι συνδεδεμένο. ο κύριο Γκουσμάου από την ΚΟΕ. Ούτε εκείνο είναι συνδεδεμένο. Κύριε εκόσα από το ΕΛΚ, και στο στο λόγο. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, λυπούμε που έχουμε τόσο πολύ απόϊχο. Η κυρία Λάγκεν Ζήπερ ε, συνδέθηκε. Η κυρία Κώσσα θα πάρει το λόγο μετά από εσάς. Η συγκήτρια νομίζω ότι έχει περάσει στο πλαίσιο της φαντασίας και θα πρέπει να επανέλθουμε στην πραγματικότητα. Το σχετικό άρθρο της συνθήκης ορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λειτουργεί. Οποιασδήποτε άλλες αρμοδιότητες είναι αρμοδιότητες των κρατών μελών. Μία από αυτές είναι η πολιτική απασχόλησης και η άλλη είναι η κοινωνική πολιτική, πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας. Κάθε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι πιστό στην αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η πληνότητα λοιπόν των τροπολογιών βάσει το άρθρου 12 έχουν να κάνουν με τον κατώτατο μισθό. Το κείμενο αντιφάσκει με τους κανόνες που έχουμε εγκρίνει και υπάρχουν τροπολογίες βάσει το άρθρου 12. Συμφωνώ με την ε, Σουηδέζα συνάδελφο που ζήτησε τη διαγραφή της παραγράφου 12. Να επισημάνω εδώ ότι η συνθήκη αναφέρει ξεκάθαρα ότι τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν το ευρώ για διαφορετικές κατηγορίες του πληθυσμού Ε, εντάσσονται σε μια άλλη καταγραφή των στοιχείων τους. Βλέπουμε εδώ να υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ μελών της Ευρωζώνης και, μελών και κρατών που δεν είναι μέλη. Αυτή η διαφοροποιημένη προσέγγιση πιστεύω αντιφάσκει με τις επιταγές της ε, συνθήκης. Συνάδελφοι λοιπόν θα σας παρακαλέσω να μην υποστηρίξετε όλα αυτά τα σημεία του κειμένου ε, και τις παραγράφους που αντιφάσκουν με το πνεύμα της συνθήκης και του Ευρωκοινοβουλίου. Ας προφυλάξουμε την εικόνα του κοινοβουλίου μας και να φροντίσουμε ο επαγγελματισμός μας να παρακολουθεί το πώς εξελίσσεται η νομοθεσία και οι κανονισμοί. Είναι στιγμή να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Κώσα. Η εισηγήτρια θα αντιδράσει μετά στις παρατηρήσεις σας και τώρα η κυρία Λάγεν που βλέπω ότι είναι συνδεδεμένη. Καλημέρα σας. Με ακούτε, με ακούτε πρόεδρε. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα συνάδελφοι. Ελπίζω να είχατε όλοι ένα καλό Σαββατοκυριακό. Θα μιλήσω εκ μέρους του συναδέλφου, της συναδέλφου κύρα Μαρή Πίτερ Χάντζεν που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα το πρωί. Κυρία Ντόμπρεφ, Ευχαριστούμε για την εξαιρετική έκθεση με την ε, πολύ καλή ε, εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε άριστα αποτελέσματα. Ως προς την οικονομία και την κρίση που διανύουμε τώρα, και εμείς ε, θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μια καλή ε, πολιτική σε αυτό το εξάμεινο για καλύτερη κοινωνική προστασία. Σε αυτό το πλαίσιο κρίσης πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να έχουν, κανονικ... να έχουν ε, θετικές συνθήκες διαβίωσης. Γι' αυτό πρέπει να ζητήσουμε μέσα από την έκθεση αυτή ένα ικανοποιητικό ελάχιστο εισόδημα. Πρέπει να τονιστεί ότι θα πρέπει να προστατευτούν οι περισσότερο ευπαθείς ομάδες Ιδίω όσοι έχουν μείνει άνεργοι λόγω της κρίσης. Οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα θεμέλια της καθημερινότητάς τους. Δεν πρέπει να τους παραβλέψουμε, ούτε να τους ξεχάσουμε στην προσπάθεια ανάκαμψης. Ίσα ίσα θα χρειαστούν περισσότερη υποστήριξη. Ε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Λάγκεν Και τώρα ο λόγος στην εισηγήτρια, κυρία Ντόμπρεφ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και μάλιστα καυτή. Ε, θα ξεκινήσουμε τις συνεδριάσεις των εισηγητών κατευθείαν μετά τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλια, για να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Είναι σημαντικό για όλους μας, γιατί όπως έδειξε και η κρίση της ε, πανδημίας του COVID-19, θα πρέπει να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη, μάλιστα να τα ενθαρρύνουμε, να επενδύσουν στο κοινωνικό σκέλος, ε, προστατεύοντας ε, τα δημόσια κονδύλια και ακολουθώντας το δρόμο της βιωσιμότητας, διότι αυτή είναι ο μόνος δρόμος και είναι σαφές ότι θα πρέπει να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη από κοινού σε όλες τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου. Από την άλλη, βλέπω να υπάρχει πολλή υποστήριξη για ε, να υπάρχουν ισχυρές ευρωπαϊκές κοινωνικές πολιτικές και χαίρομαι που η κυρία Ούρσουλα Φόντε Λάιεν αλλά και οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές και το ΕΛΚ μιλούν για κοινωνική προστασία, μιλούν για ε, κατώτατους μισθούς. Εκεί πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε κάποιο περιθώριο συνεννόησης. Άκουσα για διακρίσεις και διαφοροποίηση κρατών Ευρωζώνης και εκτός Ευρωζώνης. Να θυμίσω σε όλους μας ότι το ευρώ ε, είναι υποχρέωση όλων των χωρών που δέχτηκαν να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης. Υπάρχουν ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν εφόσον έχει εγκρίνει κανείς το κοινό νόμισμα, αλλά πιστεύω ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης θέλουν συμμετοχή στην Ευρωζώνη και ό,τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη είναι καθοριστική σημασία και για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει κοινωνικότερη, πρασινότερη, ψηφιακότερη ε, προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ιδίως στην Ευρωζώνη ε, και μάλιστα με τη διάσταση της αλληλεγγύης. Αυτό είναι σημαντικό για όλους μας και για το μέλλον μας. Προσβλέπω στη συνεργασία με τους κοιόδης Ευχαριστώ για την πληθώρα σχολείων και πιστεύω ότι θα έχουμε μια παραγωγική συζήτηση και συνεδρίαση σπιωδών. Ευχαριστούμε κυρία Ντόμπρεφ. Η ψηφοφορία θα γίνει στην ΕΜΠΛ ε, την 1η ε, Οκτωβρίου. Αυτά για τη σημερινή συνεδρίαση. Αγαπητοί συναδέλφοι, θα τα πούμε το απόγευμα στις 2 παρατέταρτο. Καλό μεσημέρι.